Dear President, Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε και ο Γενικός μας ο Κλάους Βέλε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Βρισκόμαστε εδώ για μια εξαιρετικού χαρακτήρα εκδήλωση, γιατί σήμερα πρόκειται να υπογράψουμε την ε, περιβαλλοντική ε, συνθήκη για το 2016, για το EMAS, Eco Management and Audit Scheme στα αγγλικά που είναι ένα εργαλείο διαχείρισης προαιρετικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόκειται για ένα κρογωνίο λίθο στο σύστημα ε, χείρισης του Κοινοβουλίου και η πρώτη μας τέτοια περιβαλλοντική πολιτική υπογράφεται το 2007. Από τότε δε το Κοινοβούλιο έχει ε, βελτιώσει τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις σημαντικά και η νέα πολιτική του 2016, η οποία σήμερα πρόκειται να ε, μονογραφηθεί, θα είναι μια βελτίωση ε, της προηγούμενης εκδοχής, θα είναι πιο φιλόδοξη, γιατί το Κοινοβούλιο έχει ρόλο πολύ σημαντικό όσον αφορά την πολιτική πολιτική στην Ευρώπη και για αυτό και πασχίζει για ένα βιώσιμο ε, μέλλον και εμείς στην Επιτροπή μας βέβαια είμαστε στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Η περιβαλλοντική μας πολιτική 2016 αντιπροσωπεύει το πόσο δεσμεύεται το Κοινοβούλιο το οποίο να μπορέσει να πετύχει αυτήν την βιωσιμότητα στην καθημερινή του λειτουργία. Οπότε και ε, βεβαίω είναι λογικό εμεί σήμερα να φιλοξενήσουμε την διαδικασία αυτή τη μονογράφηση τη ε, Ήμας. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Λαβία, αγαπητοί συνάδελφε της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα μαζί με εσάς ε, σήμερα να μπορώ να υπογράψω αυτό το πολύ σημαντικό έγγραφο. Επίσης, συμμερίζομαι τη δήλωση του Προέδρου, του κυρίου Λαβία, και ήθελα και εγώ να πω ότι εμείς ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε την υποχρέωση ως νομοθέτες ε, οι ίδιοι να παίξουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Να πάμε πέρα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της αλλαγής του κλίματος ως νομοθετικό όργανο και ως θεσμικό όργανο το οποίο λογικά πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι άλλοι απαιτούν από εμά νομοθεσία. Εμείς ε, φυσικά, όπως λένε όλοι, πρέπει να δείχνουμε το καλό παράδειγμα και αυτό είναι και το βασικό στοιχείο της προηγούμενης πολιτικής. Εμείς ως νομοθέτες, ως πολιτική αρχή, ως ε, διοικητική αρχή επίσης, έχουμε εδώ 8.000 ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε διάφορες ε, θέσεις και ε, καταναλώνουν ε, νερό, έγγραφα, χαρτί δηλαδή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο αποδοτικοί και να λαμβάνουμε καινοτόμα μέτρα για την διαχείριση των κτηρίων μας έτσι ώστε να φροντίζουμε το περιβάλλον οι ίδιοι πρώτα. Αυτό ακριβώς είναι και ο στόχος, ο στόχος ε, της ε, συμφωνίας που εδώ σήμερα υπογράφονται. Οι ομάδες εργασίας έχουν και διοικητική και πολιτική αποστολή. Έχουμε τη Γενική Διεύθυνση, ε, η οποία διαθέτει οριζόντιες ομάδες εργασίας που συνεχώς ε, προσπαθούν ε, να εκπληρώσουν ακριβώς αυτά τα καθήκοντα και είναι και αυτό η αρμοδιότητα του Γενικού η Γραμματέα του κ. Βέλε. Επίσης έχουμε την ομάδα εργασίας του Προεδρείου, η οποία ασχολείται κυρίως με τη διαχείριση των κτηρίων με την άμεση διαχείριση των υποδομών γενικότερα. Έχει ακριβώς αυτό το καθήκον. Ε, είναι ε, κάπως πιο περιορισμένη η εργασία του σε σχέση με την ε, διοίκηση και την πολιτική πλευρά των αποφάσεων που λαμβάνει. Εδώ όμως, ε, ως εκπρόσωποι αυτής της ομάδας εργασίας και ως πολιτικοί, ακριβώς ε, πρέπει να αναλύσουμε αυτό που μας προτείνει η διοίκηση και ε, εντατικά μεταξύ μας να κάτσουμε σε ευρύτερο πεδίο, όχι μόνο στο επίπεδο του Προεδρείου, έτσι ώστε να προσυπογράψουμε αυτό που ομόφωνα υπέγραψε το Προεδρείο κάτι που μας δεσμεύει για τα επόμενα χρόνια. Είναι μια λοιπόν πολύ καλή ευκαιρία που σήμερα ενώπιον ημών βρισκόμαστε εδώ ε, και έχουμε εσάς ως μάρτυρες ε, και ε, όλοι μαζί μπορούμε να υπογράψουμε αυτό το έγγραφο. Ευχαριστώ. Τώρα μπορούμε να κατέβουμε για την υπογραφή. Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι της συνεδρίασης και ξαναξεκινάμε στις 3.30. Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Να θυμίσω σε όλους τους συναδέλφους να χρησιμοποιήσουν την κάρτα για την ψηφοφορία, εάν χρειαστεί. Πάμε λοιπόν στο σημείο 10 της ημέρησιας διάταξης Πρόκειται για τη διατύπωση αντιρρήσεων ε, σύμφωνα με το άρθρο 106. Ανώτατα όρια καταλήπων για την ουσία τριακλοπρίντ μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. Λοιπόν, υπάρχει ένα αίτημα από την εισηγήτρια να ψηφίσουμε ονομαστικά για, αυτήν την, για αυτό το ψήφισμα. Θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχουν 17 μέλη που να είναι υπέρ της ονομαστικής πλειοψηφίας, ε, ψηφοφορία, συγγνώμη. Λοιπόν, πώς είναι υπέρ. Everybody voted. Μάλιστα, ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Mr. Pedicini, how have you have voted? Yes, but you... Ψηφίσατε. Ψηφίσατε υπέρ, κατά, υπέρ. Μάλιστα. Μάλιστα. Ψηφίζουμε λοιπόν με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Για η διατύπωση αντιρρήσεων. Πέρας της ψηφοφορίας, συν τον κύριο Πεντητσίνη. Λοιπόν, η διατύπωση αντιρρήσεων απορρίπτεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε για το σημείο 11 Πρόκειται για την εντολή για την έναρξη του τριμερούς διαλόγου για τον προπολογισμό του 2017. Ξεκινάμε με την τροπολογία 1. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα να ψηφίσουμε την τροπολογία υπερθυμών 6 η οποία είναι συμβατή. Ψηφίζουμε την 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η επόμενη υπέρ κατά εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε την τροπολογία 17 του συναδέλφου κάπου το υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε την 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 σε δύο τμήματα το πρώτο υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος ψήφισαν όλοι πέρας εγκρίνεται Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία 23 σε δύο τμήματα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Τελική ψηφορία ηλεκτρονικά. Συγγνώμη, συγγνώμη και ο πρόεδρος. Τώρα ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στο 12. Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέρμανση και την ψήξη. Votiamo il compromesso 1. Φιέλνερ, ο συγκητής, πρώτη συμβαστική υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8, υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος ψήφισαν όλοι Πέρασε. Εγκρίνεται. Πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα συμβαστική εννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη. Και τώρα ψηφίζουμε την επτά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψήφισαν όλοι πέρας. Έγκρινε. 24 υπέρ. Κατά. Άποχη. Εγκρίνεται. Το 25 υπέρ. Κατά. 26, 26, συγγνώμη, συγγνώμη. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία για την τροπολογία. 26, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 σε δύο τμήματα το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεν ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα, οπότε πάμε στο 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψήφισαν όλοι. Πέρασα. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 34. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε το 41 σε δύο τμήματα όχι όχι όχι όλο μαζί όλο μαζί το κείμενο της 41 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβεστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Συνδεθεί δέκα υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 σε δύο τμήματα. Το πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψήφισαν όλοι, πέρασε. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την ε, τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπερθυμών 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Και εγκρίνεται. Εμενταμέντο 63. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω, αλλά ας γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4α. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψήφισμε την τροπολογία 73. È compatibile come un'aggiunta al compromesso. Ε, συμβατό αυτό ως προσθήκη στο 4α. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε το 73. 73. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Ιδρυτικός έλεγχος. Avete votato tutti? Ψήφισαν όλοι. πέρα Και εγκρίνεται. Και τώρα η 76. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. 77 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψήφισαν όλα, πέρας. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το 84. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα ψηφίζουμε το 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 υπέρ Κατά. Α, αποχές. Έλεγχος. Περίεργη πλειοψηφία. Ψήφισαν όλοι. Και εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι, πέρας και εγκρίνεται. And now We can go to 13 in our agenda, uh, the vote on... Και τώρα περνάμε στο σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης. Ε, θα μιλήσει η συγγήτρια σχετικά με το θέμα της επικορικότητας. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα, θα ήθελα να διατηρήσω ε, τις λύσει λύσεις και χαίρομαι που το ΕΛΚ είναι το, η, μόνη, η πολιτική παράταξη που μας υποστήριξε. Εδώ υπάρχουν ε, συμβαστικές προτάσεις από όλα τα κόμματα και από τους φιλελεύθερους ε, και από τους πράσινους και από το ΕΛΚ θα ήθελα να ψηφιστούν από την αρχή οι συμβαστικές προτάσεις με ονομαστική ψηφοφορία. Να πω επίσης ότι πολλές από αυτές τις τροπολογίες ήρθαν να εμπλουτίσουν το κείμενο και δεν υπήρχε κάποια ουσιαστική αντιπαράθεση εκτός από κάποιες περιπτώσεις που ήδη όμως αφαιρέθηκαν στην αρχική εκδοχή του συμβασμού. Δεν άκουσα κανένα επιχείρημα ουσίας όμως ε, που να οδηγεί σε αντιπαράθεση. Κάποιες ομάδες ζήτησαν να βγουν από τις συμβαστικές λύσεις χωρίς να εξηγήσουν το γιατί, ενώ τα κείμενα αυτά λάβαναν υπόψη τα επιχειρήματά τους και των τροπολογιών τους. Επίσης το κόμμα ECD έχει αποσύρει όλες τις τροπολογίες του χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Λυπάμαι που παρότι εμείς την, ανοίξαμε τα χέρια μας, ε, υποστηρίξαμε νομοθετικές πρωτοβουλίες συναδέλφων και στο παρελθόν, μόνο και μόνο η πολιτική μου ε, στράτευση ε, προκάλεσε ε, απόρριψη χωρίς επιχειρηματολογία και αυτή η στάση απέναντι σε μένα προσωπικά και στο κόμμα μου, στην ομάδα μου, ε, είναι πραγματικά ατιμωτική το να διατηρά, διατηρείται αυτήν την τεχνητή ε, αντιπαράθεση είναι δηλητήριο για τις κοινωνίες μας. Μάλιστα. Συνάδελφοι, να μην ξεκινήσουμε συζήτηση για αυτό το θέμα. Είχε το λόγο η συγγήτρια και ζητήθηκε νομαστική ψηφοφορία για το συμβιβασμό. Ρώτησαν υπάρχουν 17 υπέρ της ονομαστικής. Ελπίζω ότι ε, αν είμαστε υπέρ θα, ψη, θα υπερψηφιστεί. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Everybody voted. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορία. 15 υπέρ και θα ψηφίσουμε χωρίς να έχουμε νομοριστική ψηφοφορία. Εμενταμέντο 9. υπερθμό είναι 9 που είναι υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Λειτουργικός έλεγχος. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13. Έχει αποσυρθεί. Πρέπει να ψηφίσουμε το 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Α, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Α, αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το 17 υπέρ. Κατά. Α, αποχές εγκρίνεται. 18. Καταπίπτει. Πάμε στο 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Παρακαλώ να σηκώνετε σαφώς τα χέρια σας, συνάδελφοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. πρέπει να ψηφίσουμε το 20 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Κατά πίπτη και ψηφίσουμε την τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τοπολογία 23. Είναι γλωσσικού χαρακτήρα. Α, όχι, όχι. Πρέπει να το ψηφίσουμε, μου λέει η γραμματεία Το 23, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3. Συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 σε δύο τμήματα. Το πρώτο περ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 δύο τμήματα. Πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 32 υπέρ κατά Α, αποχές απορρίπτονται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψήφισαν όλοι πέρας, εγκρίνεται. Και τώρα ψήφισαν το 41 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Ingrid. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτονται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πενήντα ένα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτωτο. 52 υπέρ. Κατά. αποχές απορρίπτωτο. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτωτο. Περιθμόν 1 υπέρ. Κατά. Α, αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει το 2 και πάμε στο 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική παριθμών 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. We have finished to vote. Ολοκληρώσαμε την ψηφοφορία. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην μέση διάταξη. Καλό λοιπόν όλα τα μέλη τα οποία ε, εγκαταλείπουν την αίθουσα να το κάνουν γρήγορα. Γιατί πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Το επόμενο σημείο στην ημέρησα διάταξη είναι η ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με τα κριτήρια βιωσιμότητας για τη βιομάζα. Μόλις οι συνάδελφοι αποχωρήσουν, θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ακούσουμε τη θέση της και να ξεκινήσει η ανταλλαγή απόψεων. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ αποχωρήστε ησύχως και ταχαίως. Ο κύριος Πίτερ Άντλεϊ έχει το λόγο από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που θα μας παρουσιάσει τη θέση της Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ, εκ μέρου του Ζωάν Ερικ Πακέ που σκόπευε να έρθει σήμερα διότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα για την Επιτροπή σας. Δυστυχώς ε, ε στην Επιτροπή του από το Άμστερνταμ κάπου ε, έμπλεξε, κάπου κόλλησε και ήρθα εγώ. Αντί γι' αυτό Θέλω να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή Περιβάλλοντος που οργανώνει αυτή την ανταλλαγή απόψεων η οποία έρχεται, λαμβάνει χώρα μια κέρια, σε μια κέρια χρονική στιγμή, καθώς εξετάζουμε την ανάλυση που θα οδηγήσει σε μια πρόταση, πολιτική πρόταση για την ε, βιωσιμότητα της βιοενέργειας. Ε, έχω εδώ συναδέλφους από όλε τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εμπλέκονται στην προπαρασκευή αυτής της πολιτικής. Αυτό δείχνει ότι έχει πολλές ε, πολλούς τομείς ε, που επηρεάζονται, περιβάλλον, ε, γεωργία, εμπόριο. Η βιοενέργεια δεν είναι μια πολιτική αυτόνομη. Ε, η γνωμοδότηση που μόλις εγκρίνατε για την θέρμανση και την ψήξη, εκεί η βιοενέργεια και, ήδη, και ιδιαίτερα η βιομάζα μπορεί να συνεισφέρουν σημαντικά. Επίσης συνδέεται και με τις προτάσεις για το κλίμα που θα υποβάλει η Κομισιόν πριν από το καλοκαίρι για την αλλαγή της χρήσης της γης, της εντομέρειας δασοκομείας και την κατανομή της προσπάθειας. Θα γίνουν και προτάσεις, προτάσεις μετά το καλοκαίρι για την ε, αποδοτική χρήση της ενέργειας, καθώς και αργότερα φέτος για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και βεβαίως ε, το θέμα του σχεδιασμού της αγοράς λειτουργικής ενέργειας και το σχεδιασμό της Ενεργειακής Ένωσης συνδέεται επίσης με ευρύτερες πολιτικές ανησυχίες, οι ε, στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη και οι στόχοι που παρουσίασε η Κομισιόν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Προετοιμάζουμε την πολιτική μας πρόταση αυτή τη στιγμή. Νωρίτερα φέτος έλαβε χώρα μια δημόσια διαβούλευση όπου συμμετείχαν πάνω από χίλια, είχαν πάνω από χίλιες απαντήσεις μάλλον και στις 10 Μαΐου είχαμε και μια συνάντηση των εμπλεκομένων φορέων, έγιναν πολλές μελέτες και έχουμε πλέον, ε, συμπτήσουμε τα στοιχεία στα οποία θα βαστεί η πολιτική μας, εμείς θα σεβαστούμε απολύτως τις αρχές της καλής νομοθεσίας. Το πρώτο ερώτημα που θέτουμε είναι γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για την βιώσιμη βιοενέργεια. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι βασιζόμαστε στη βιοενέργεια ε, δύο τρίτα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που που ε, παράγονται στην Ευρώπη προέρχονται από την βιοενέργεια. Έχουμε ήδη μια πολιτική βιωσιμότητα για τα βιοκαύσιμα, αλλά δεν έχουμε μια τέτοια πολιτική για τη βιομάζα. Και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για, το πλαίσιο, για το κλίμα και την ενέργεια του 2030, είπαμε ακριβώς ότι θα εκπονήσουμε μια τέτοια πολιτική για να, να συνοδεύσει τους στόχους που έχουμε θέσει για το 2030. Ε, να σας πω έτσι εν συντομία τι είδου ζητήματα εξετάζουμε. Πρώτα απ' όλα εξετάζουμε ποια είναι η συνεισφορά της βιοενέργειας στη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Δεύτερον, εξετάζουμε το περιβαλλοντικό αντίκτυπο της χρήσης της βιοενέργειας, το θέμα της βιοποικιλότητας, της ε, ρήπανσης της ατμοσφαιρικής, της ε, ρήπανσης των ε, υδάτων, της γης, Εξετάσαμε επίσης το κατά πόσο είναι συμβατά αυτά με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Επίσης εξετάζουμε την οικονομική και κοινωνική διάσταση του ζητήματος. Ιδιαίτερα τη διαθεσιμότητα βιομάζας ε, από τα δάση για να μπορέσει να στηριχθεί αυτή η πολιτική στο μέλλον και για σκοπούς που δεν έχουν σχέση με την ενέργεια. Εξετάζουμε ποια, σχέση, ποια θέση παίρνει η πολιτική της βιοενέργειας ε, για την, ανάπτυξη, στην απασχόληση, στην ανάπτυξη της υπαίθρου και στις κοινωνικές προσαρμογές. Τέλος, εξετάζουμε τη βιοενέργεια σε ό,τι αφορά τα θετήματα της ενεργειακής ασφάλειας, διότι άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, ε, μπορεί να είναι μεταβλητές, όπως ο ήλιος και ο αέρας, εδώ όμως δεν είναι η περίπτωση. Ε, αυτή. Εξετάζομαι τα διάφορα ζητήματα λοιπόν. Δεν είναι ακόμα, δεν είμαστε έτοιμοι να σας πούμε ποιες είναι οι εναλλακτικέ τις οποίες ε, καταλήγουμε ή ποιο νομοθετικό μέσο θα επιλέξουμε αργότερα φέτος, αλλά καλό θα είναι να έχουμε την άποψη της Επιτροπής για τα ζητήματα αυτά. Σκοπεύουμε να βασιστούμε σε ε, στοιχεία επιστημονικά αξιόπιστα και να ε, ε, σεβαστούμε απολύτω τι αρχέ τη αναλογικότητα και τη επικουρικότητα. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε περιβολικό διοικητικό άρθρο για του οικονομικού φορεί, ούτε να εμπλακούμε σε τομεί όπου η αρμοδιότητα είναι των κρατών μελών. Θα σεβαστούμε επίση του διεθνεί κανόνε ε, για το εμπόριο και θα εξασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε πολιτική επιλέξουμε ε, θα συνεισφέρει για τη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, όπως άλλωστε αναφέρεται στι δεσμεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της Συμφωνίας του Παρισιού. Αναμένουμε λοιπόν αποτελέσματα ρεαλιστικά, ισορροπημένα, συνεκτικά και συνεπή με άλλε πολιτικές τη Ένωση και κυρίως στέρεα. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, αναμένουμε μια επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ξεκινάμε Ξεκινάω άμεσα με ένα ερώτημα στα Ιταλικά. Ε, Υπάρχει μεγάλη ευρωπή στην Ευρώπη, οπότε έχουμε και κάποια μέτρα τα οποία είναι δυνατόν να μπορέσουν να θεσπιστούν και έχουμε και κάποια άλλα κριτήρια της βιωσιμότητας τα μπορούσαν μπορούμε να μετέλθουμε όσον αφορά τα δάση και την ε, βιομάζα και αυτό ιδιαίτερη σημασία έχει για τον Νότο. Και όταν δε μιλούμε για το ΆΕΛΟΚ ως μεταβλητήριο παράγοντα έχουμε λάβει υπόψη κάποιες κυκλικές μεταβολές που θα μπορούσαν να γίνουν παραδεκτές και επομένως ίσως δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Όμως έχουμε ακόμα εκατομμύρια εκταρίων γιατί έχουμε αυτού του είδους την κυκλική εναλλαγή στις καλλιέργειες. Οπότε έχουμε αυτή την αγρανάπαυση των οσέδους, οπότε και έτσι ε, υπάρχει εξοικονόμηση υδάτων για την επόμενη χρονιά. Όμως ε, αυτή η πρακτική αντέχει στον χρόνο, γιατί όταν χρησιμοποιούμε για κάποιο είδους βελτιωτικές καλλιέργειες το έδαφος, τότε αυτό θα φέρει μια επιδείνωση όσον αφορά το νερό ή τον υδροφόρο ορίζοντα και αυτό θα έχει επιπτώσει για την επόμενη χρονιά. Οπότε θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι η καλλιέργεια κάποιων ειδών που δεν αντιστοιχούν σε κάποια αγορά αλλά θα μπορούσαν να βοηθήσουν για την παραγωγή βιομάζας επίσης βοηθούν στην απορρόφηση του διοξιδίου του άνθρακος από την ατμόσφαιρα και επίσης μπορούμε σε κάποιες ζώνες να έχουμε κάποια στοιχεία οργανικά τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην βιωσιμότητα που θέλουμε. Ένα άλλο κριτήριο αυτό. Και έτσι να έχουμε τέτοιου είδους ε, παραγωγή που μπορεί να μην έχει να μην σε κάποια αγορά αλλά αυτό ισχύει να και κάποιες ε, ζωοτροφές. Οπότε αυτές οι φορτοκαλλιέργειες έτσι κι αλλιώς βοηθούν στο να έχουμε περισσότερο πράσινο υλικό το οποίο να, μετά την ορίμανσή του να βοηθά και να αποτελεί ύλη, πρώτη ύλη για παραγωγή βιοαερίου. Κύριε Ριβαζίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στα κριτήρια της ε, διάρκειας και να σας δείξω ένα παράδειγμα που γίνεται στην Μασαλία, στο Περκαρντάνο, όπου υπάρχει ένα θερμικό εργοστάσιο που χρησιμοποιεί 800 ε, ε, εκατομμύρια τόνους για να παράγει ηλεκτρισμό. Λέτε ότι θέλουμε να μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου, όμω το περισσότερο ξύλο που χρησιμοποιείται στις, στη Μασαλία έρχεται από τον Καναδά. Αυτό είναι ένα κριτήριο που πρέπει να ε, έχουμε για να μπορέσουμε να απαγορεύσουμε τη μεταφορά ξυλίας από τον Καναδά στη Μασαλία. Ποιο είναι αυτό, ε, να μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου. Μόνο και μόνο για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Λοιπόν, ε, να μην χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτή την θερμότητα που παράγει το θερμικό εργοστάσιο. Θεωρώ λοιπόν ότι η ενεργειακή ε, αποδοτικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική και υπάρχει και ένα κείμενο που ουσιαστικά απαγορεύει αυτού του είδου τη βιομηχανία. Ότι ε, φαίνεται ότι τα γειτονικά δάση πάσχουν επειδή ε, και όλα κόβονται γιατί χρησιμοποιούνται ε, για αυτό τα εργοστάσια. Επίσης καταδικάζει και το κλίμα αλλά και τις Ε, όλα αυτά τα, ε, όλες αυτές τις συσκευές που χρησιμοποιούν την ξυλία για, την, ε, για να θερμάνουν το νερό. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη ένταση σχετικά με αυτή την απαγόρευση της μεταφοράς ξυλίας από τον Καναδά. Ήθελα να πω και εγώ όμως κάτι που είπε ήδη ο Πρόεδρος. Έχουμε ήδη κάνει μία συζήτηση με τον Επιτρόπο στην Επιτροπή ε, Γεωργίας σχετικά με τη ε, κριτήρια για την βιομάζα και φαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρυσι ε, είχε ψηφίσει μία έκθεση, μία στρατηγική η οποία μιλούσε ακριβώς ε, για την ε, ε, βιώσιμη διαχείριση στην Ευρώπη, διότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος θόρυβος για αυτό το θέμα, πάρα πολλές φωνές στην Ευρώπη που μιλούν για αυτήν την βιώσιμη διαχείριση στην Ευρώπη. Ενδιαφερόμαστε λοιπόν ε, να έχουμε αποτελέσματα τα οποία ε, θα βοηθούν τους ανθρώπους στις διάφορες περιφέρειες και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τάχθηκε ξεκάθαρα κατά των νέων κριτηρίων για τη βιομάζα. Είναι ένα θέμα βέβαια αυτό, διότι έχουμε ήδη τέτοια κριτήρια βιωσιμότητα στην Ευρώπη. Απλώς τώρα ε, είναι η πρώτη φορά που πρέπει να ψηφίσουμε κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν και με τα δάση. Υπάρχουν κριτήρια, δεν είναι όμως ε, πιο ε, στοχευμένα και να λένε πώς θα αντιμετωπίσουν διάφορες περιφέρειες στα δάση έτσι ώστε να μην υπάρχει αλλαγή του κλίματος και ποια είναι η κοινωνική επέκταση του θέματος. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Κομισιόν αν ε, ξέρει αυτή την ε, θέση του Κοινοβουλίου ε, και αν θα ληφθεί υπόψη αυτή η θέση. Ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Φίλνερ. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχηθώ καλή τύχη στην Επιτροπή για αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο ζήτημα. Ε, είναι γεμάτος παγίδες ο δρόμος, ο δρόμος όμως προς την κόλαση φαίνεται ότι έχει στρωθεί με καλές προθέσεις. Όπως και να έχει, η φιλοδοξία είναι μεγάλη. Έχω τρία ερωτήματα. Με μεγάλη μου χαρά άκουσα την Κομισιόν να λέει ότι ήταν πολύ προσεκτική όταν τέθηκε το θέμα της επικουρικότητας, κυρίως επειδή ε, το θέμα το δασικό δεν είναι στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν σχετίζεται με τα κριτήρια της βιωσιμότητας. Είναι δύσκολο κανείς να ασχοληθεί με τη βιωσιμότητα χωρίς να μιλήσει για τα δάση. Οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι το είχαν σκεφτεί αυτό, γιατί ε, εδώ, σε αυτή την αίθουσα, αν είχαμε κάνει, ανοίξει τη συζήτηση ακόμα και για τον ορισμό του δάσου, θα είχαμε διαφωνήσει. Ε, όταν η Φιλανδία και η Σουηδία μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1995, κατά 50% αυξήθηκαν οι δασικές εκτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είναι λάθος λοιπόν ε, αυτό, υπάρχει τεράστια αντίδραση που θα προκύψει από αυτές τις χώρες. Άρα, ερώτηση, πώς είναι δυνατόν να ρυθμίσουμε τα βιώσιμα κριτήρια χωρίς ε, να ρυθμίσουμε τη διαχείριση των δασών που δεν είναι στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, ένα άλλο ε, πολύ σημαντικό ερώτημα που πρέπει να το σκεφτούμε πολύ πριν ε, ασχοληθούμε με το οδηγία των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια είναι η σχετική ανταγωνιστικότητα των πηγών αυτών, γιατί δεν έχουμε κανένα κριτήριο βιωσιμότητας για τα ορυκτά καύσιμα, τον άνθρακα, το αέριο. Έτσι, λοιπόν, αν ενισχύσουμε τα, στριχή, τα κριτήρια βιωσιμότητας για τα πράγματα που μας αρέσουν, επειδή μας αρέσουν, θα τα σφίξουμε τόσο σφιχτά στην αγκαλιά μας που θα τα πνίξουμε. Ε, νομίζω, λοιπόν, ότι ε, αυτό ε, είναι πολύ σημαντικό. Τι μπορούμε να πούμε, βέβαια, για τη βιομάζα. Ε, όταν υπάρχουν παραδείγματα που μπορεί κανείς να βρει ε, που θα ισχυρίζονται ότι είναι χειρότερο από το άνθρακα. Ε, όμως, αν κάνουμε κάτι, και αυτό δεν είναι θεωρητική σκέψη, τα κλαδάκια και τα κολοβόμετα που θα μείνουν έξω εκεί έξω ε, δεν θα είναι βιώσιμα γιατί δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Η δική μου εμπειρία δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολο κανείς να φτιάξει νομοθεσία και να δούμε πώς ε, θα ορίσουμε το πώς θα χρησιμοποιεί ο καθένας το οτιδήποτε. Η διαδικασία διαδοχικών σταδίων είναι πολύ δύσκολη θα έλεγα θεώρησα λοιπόν ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να μην χρησιμοποιήσει μια τέτοια διαδικασία γιατί είναι κομμάτι ενός επιχειρηματικού μοντέλου. Αν το κάνουμε νόμο, θα καταλήξουμε με μια σχεδιασμένη οικονομία που δεν λειτουργεί. Θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να ακούσουμε τα σχόλιά τους γι' αυτό. Thank Ευχαριστώ, κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ ε, ήθελα να συνεχίσω ε, αυτή τη συζήτηση διότι την παρακολουθώ εδώ και πολύ καιρό. Ε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δω και να κατανοήσω τις διάφορες μορφές βιομάζας διότι είναι πολύ σημαντικά για πολλά ζητήματα. Το 46% της βιομάζας είναι ε, το, ε, η ξυλία ξεκάθαρα. Η ε, βιωσιμότητα είναι ένα κομμάτι της διαχείρισης των δασών και πρέπει αυτή η διαχείριση να είναι ενεργή και πρακτική, πρακτικά να τη χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα δάση. Έχουμε στο μεταξύ ε, τους δύο ε, τα δύο σήματα που ε, διασφαλίζουν ότι έχουμε μία βιώσιμη διαχείριση των δασών. Ε, αυτό πρέπει να το έχουμε στις εισαγωγές ξυλίας για να μπορούμε να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της δικής μας δασικής οικονομίας. Ε, πρέπει αυτά που εισάγουμε να, να υπακούν στις ίδιες αρχές με αυτά που παράγουμε εδώ στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε, να μην έχουμε εδώ επιπλέον κριτήρια με επιπλέον γραφειοκρατία που θα ε, δημιουργήσουν προσκόμματα στη δική μας δασική ε, οικονομία. Ε, θα πρέπει να πω ότι ο τομέας αυτός ανήκει στην ευθύνη των κρατών μελών. Δεν θέλουμε να υπάρξει ε, κάποια μεταφορά των αρμοδιοτήτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και επέκταση αυτών. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί οι καλύτεροι εγγυητές ε, της βιωσιμότητας της ε, οικονομίας αυτής είναι αυτοί που στην καθημερινή τους πρακτική ασχολούνται με το ζήτημα και δουλεύουν γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριο Πεντησίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ Θέλω να σας μιλήσω για το ότι τελικά ό,τι κριτήριο και να επιλέξουμε βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλούς πρώιμους θανάτους λόγω των ουσιών που δημιουργούνται από αυτές τις καλλιέργειες και από την παραγωγή της βιομάζας. Το ίδιο ε, γίνεται και με την διοξίνη Οπότε έχουμε διάφορες εκπομπές που προέρχονται και από τα αυτοκίνητα ή τέλος πάντων από τη διαδικασία παραγωγής της βιομάζας. Έχουμε συζητήσει ήδη αυτό όταν ζητούσαμε την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και είπαμε ότι θέλουμε να καλύψουμε την περίοδο από το 2020. Και έχουμε τις ε, συστάσεις προς τα κράτη-μέλη που ξέρουμε όμως ότι δεν θα εφαρμοστούν. Θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα δεσμευτικά και θαραλέα. Είχαμε ένα εργοστάσιο στην Νότια Ιταλία από το 1962 και παρά τις διαδικασίες για χορήγηση έγκρισης τελικά τίποτα δεν έγινε και χρησιμοποιούνται κάποια καύσιμα τα οποία είναι ρηπαντικά. Το 2016 έχουμε επίσης έλλειψη της έκθεσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οπότε θα πρέπει να μας απαντήσει όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί υπάρχουν τόσα κενά στο ρυθμιστικό πλέγμα και επίσης θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να συνειδητοποιηθεί ότι δικαιούνται να αναπνέουν καθαρό αέρα. Τα κριτήρια αυτά της βιωσιμότητας για την βιομάζα τα έχετε καθορίσει αλλά είπαμε ότι δεν είναι συμβατά με τον φυσιολογικό κύκλο της φύσης. Άρα αυτά είναι για το σημείο των Ευρωπαίων ή όχι. Κύριε Άουκεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ είναι ότι δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε τη φύση. Κάποιος εδώ μίλησε για τη βιομάζα και είπε ότι είναι ουδέτερη από πλευράς ε, άνθρακα. Ε, αυτό δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι αυτές οι εκπομπές δεν καταμετρούνται στην UCF όμως. Κάποιες χώρες δηλαδή αυξάνουν τις οδιές και δεν μετράμε τις αρνητικές επιπτώσεις. δεν είναι σαφής ο τρόπος καταμέτρησης από την UCF επίση. Ζητούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα επιβεβαιώσει καταρχήν ότι αναγνωρίζει τα επιστημονικά στοιχεία και αν συνεχίζει, εν πάση περιπτώσει, να χαρακτηρίζει τη βιομάζα ουδέτερη από επιστημονικής πλευράς. Τα κριτήρια βιωσιμότητα πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία για τη βιοενέργεια και πρέπει να μείνουν εκτός της βιοενέργειας ε, οποιαδήποτε μορφή η οποία οδηγεί σε αύξηση του, του άνθρακα. Ευχαριστώ κύριος Εκχάρτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το βασικό που θα ήθελα να αναφέρω εγώ είναι κατά πόσο μπορούμε να έχουμε σωστό ε, αποτέλεσμα σε λογιστικό επίπεδο. Μ' αρέσει πάντα να ακούω τον κύριο Φιέλνερ βέβαια, ιδιαίτερα όταν μιλάει για, τη, για τα δάση και τα δοσοκομεία και όταν κάνει τη σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Αφού τον αφορά τόσο πολύ το θέμα, να μένω πλήρη υποστήριξη από την πλευρά του όταν ε, προτείνουμε το τέρμα, το, το, το, τον τερματισμό των ε, επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, αλλά η ομάδα του ε, είναι κατά όταν τα συζητάμε αυτά. Κύριε Φιέλνερ, αν μπορούμε να δώσουμε αυτή τη μάχη μαζί, εγώ με ανυπομονησία το περιμένω. Σε ό,τι αφορά τώρα τη βιοενέργεια, το θέμα είναι ότι το προωθούμε αυτό με τις πολιτικές μας. Αυτή τη στιγμή προωθούμε τη βιοενέργεια. Και εφόσον το κάνουμε αυτό, πρέπει να είναι σωστά η σωστή καταμέτρηση, αν θέλετε. Και αυτό είναι που μας απασχολεί εμάς. Γίνεται σωστά η καταγραφή και αυτό είναι αρμοδιότητα της Ένωσης. Ασφαλώς και είναι ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί εδώ να μας βοηθήσει, να μας διαφωτίσει για κάποιες από τις μελέτες που, έχουν, που έχει κάνει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι σε μελέτη της Γενικής Διεθνής Ενέργειας, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στον άνθρακα για τη βιομάζα, ε, εδώ λέγεται ότι η χρήση της βιοενέργειας χωρίς όρια θα οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών της τάξης των 520 μεγατόνων. Εάν αυτό είναι ήδη το συμπέρασμα στις δικές σας εκθέσεις, Νομίζω ότι αρχίζει να γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Η Κομισιόν υποβάλλει μια πρόταση όπου θα γίνεται μια σωστή καταμέτρηση, μια σωστή προσμέτρηση. Να μας πει η Κομισιόν τι θα κάνει από αυτού. Εάν δείτε τώρα τη μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, θα, και πάλι λέγεται ότι η αύξηση της ζήτησης για βιοενέργεια θα δημιουργήσει αύξηση της χρήσης ε, του, της ξυλίας. Ε, όλοι ξέρετε ότι αν αρχίσουμε ξαφνικά να καίμε ξύλο, σίγουρα είναι αρνητικό το αποτέλεσμα για τον άνθρακα. Λοιπόν, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι για αυτό που εμείς ονομάζουμε βιοενέργεια ε, δεν θα υπάρχει κάποιος υψηλός κίνδυνος. Θα είναι χαμηλού κινδύνου βιοενέργεια αυτή ή υψηλού. Χρειάζεται, χρειάζεται λοιπόν σαφείς κανόνες για την προσμέτρηση που να ταιριάζουν τα κριτήριά μας και βεβαίως εμπίπτει απόλυτα στις αρμοδιότητες της Ένωσης. Διότι προωθούμε αυτές τις αναλλακτικές τις πολιτικές μας να το κάνουμε όμως αυτό με σωστό τρόπο και όπως είπε η κυρία Χάλγεν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε ότι η βιοενέργεια είναι ουδέτερη από πλευράς ε, παραγωγής άνθρακα, διότι δεν είναι. Ευχαριστώ η κυρία Σεργέ Πυρίκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε έχω μια διαφορετική ερώτηση να θέσω. Όταν μιλάμε για βιομάζα, η Κομισιόν πού βρίσκεται το σημείο ισορροπία τελικά. Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και στη Γερμανία χρησιμοποιείται η βιομάζα. Όμως τα φορτηγά κάνουν εκατοντάδες χιλιόμετρα για να φέρουν τη βιομάζα στις εγκαταστάσεις στις, στα, στις εγκαταστάσεις των θερμικών εργοστασίων. Και βεβαίως αυτό μπορεί να το κάνουν εύκολα οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Οι μικροί εκμεταλλευτές όμως δεν μπορούν να το κάνουν. Η βιομάζα έχει να κάνει με την παραγωγή τροφίμων, έτσι. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω κάποια περισσότερα πράγματα για τους γεωργούς εδώ. Υπάρχουν και και εθνικές. Πολείται ένα προϊόν από τους παραγωγούς διασυνοριακά. Μες στη βιομάζα περιλαμβάνουμε ε, και τα απόβλητα ορισμένε φορές ε, ε, και τα λοιπάσματα. Όμως υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία γίνονται αποδεκτά στην Ολλανδία αλλά όχι στη Γερμανία. Πρέπει να μπορεί να γίνει η, αγορά και εκτός του εθνικού επιπάδιου. Ο κ. Γκερμπάντη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε είναι κάπως περίεργη αυτή η συζήτηση. Είμαστε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, όπου συχνά βεβαίως μιλάμε για βιωσιμότητα, ε, υποστηρίζουμε τη βιωσιμότητα και ξαφνικά όταν μιλάμε για τα δάση ε, δεν μπορούμε να το συζητάμε πια αυτό. Για τα δάση η βιωσιμότητα δεν είναι θέμα συζήτησης ε, και δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν νομίζω οι ιδρυτές της Ένωσης να αποφάσισαν ε, εσκεμένα να μην συμπεριλάβουν την πολιτική δασοκομεία στο κεκτημένο της Ένωσης. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να μην συζητούμε ε, τις πρακτικές σε μικρή κλίμακα κάπου στη Βόρεια Σουηδία ή στην Αυστρία. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι με τις υφιστάμενες πολιτικές αλλά και τις μελλοντικές από ό,τι φαίνεται αυξάνουμε την χρήση της βιομάζας. Να σας πω τι γίνεται στη χώρα μου, στην Ολλανδία. Εμείς επιδοτούμε την χρήση βιομάζας. Ξύλο, έτσι, ξύλο το οποίο εισάγεται από τον Καναδά. Για να τα χρησιμοποιήσουμε στους ε, σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό το ονομάζουμε πράσινη ενέργεια και το χρειαζόμαστε αυτό για να είμαστε προτελευταίοι και όχι τελευταίοι στον κατάλογο. Ακόμα και έτσι όμως δεν τα πάμε και πολύ καλά. Δεν έχουμε καλά αποτελέσματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Εφόσον έχουμε πολιτικές οι οποίες αυξάνουν τη χρήση βιομάζας, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η βιομάζα χρησιμοποιείται κατά βιώσιμο τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζω έντονα τα κριτήρια βιωσιμότητας για τη βιομάζα. Και αυτή η Επιτροπή πάντα το έπρατε αυτό. Το ερώτημά μου τώρα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εξής. Ποια είναι η αποψή σας ε, για το co-firing της βιομάζας σε κάποια εργοστάσια. Η καύση δηλαδή ε, κάρβουνο άνθρακα. Ορισμένε φορέ έχουμε 25-40% ενώ θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό από πλευρά τη ενεργειακή αποδοτικότητα να χρησιμοποιούμε τη βιομάζα σε ειδική ε, μονάδα για την καύση βιομάζας. Δεν ξέρω αυτό το coal firing, η χρήση δηλαδή της βιομάζας ε, σε ε, εργοστάσια άνθρακα, πώς το βλέπετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι κάπως παράδοξη αυτή η ζήτηση. Εγώ προέρχομαι από κάποια χώρα που έχει μια μακρά παράδοση βιώσιμης δασοπονίας και δασοκομείας τέλο πάντων επί πολλούς αιώνε. Και οι πρώτοι νόμοι που ρύθμιζαν όλα αυτά, ξέρετε, θεσπίστηκαν, τον 14ο αιώνα. Πολύ παλιά νομοθετήματα. Ενδεχομένω, έχουμε κάποιες χώρες οι οποίες δυστυχώς ξεμπέρδεψαν με τα δάση τους. Όμως, αλλά βέβαια ο προγραμματισμός για τα δάση δεν είναι θέμα μίας κοινοβουλευτικής θητείας ή δυο ή δέκα. Είναι θέμα αιώνων. Επομένως αυτό το οποίο εγώ θέλω να σας προτείνω είναι το να είμαστε πολύ προσεκτική όποτε προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, να ρυθμίσουμε τη διαχείριση των δασών. Πάρα πολύ καλό ότι θέλουμε να νομοθετήσουμε τα της βιομάζας και τα των εισαγών από τρίτες χώρες και να εφαρμόσουμε προσεκτικά και αυστηρά τις κείμενες διατάξεις για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Όλα αυτά εντάξει σίγουρα. Αλλά, αλλά προσοχή. προσοχή να μην αρχίσουμε τα κράτη-μέλη να ανταγωνιζόμαστε σχετικά με το ποια κριτήρια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Γιατί τελικά μπορεί να καταλήξουμε να συζητούμε το ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εξάγει τελικά ο ένας τον άλλο απόβλητα και να μετακυλεί ο ένας το πρόβλημα των αποβλήτων στον άλλο. Άρα όταν κουβεντιάζουμε για τα δάση θα πρέπει να δούμε ποιες χώρες ήδη έχουν βιώσιμα δάση. Μάλιστα, μάλιστα. Λέει ο πρόεδρος, ωραία κυρία Πέτυρ, πρόεδρε, εγώ σας με θυμίζω ότι σύντομα εγκρίναμε μία έκθεση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και στο σώμα αυτής της έκθεσης αναφέρονται κάποια κριτήρια για την βιομάζα. Επίσης λέγαμε ότι θα πρέπει να λάβουμε πώς την γλυκή οικονομία και βιώσιμες πολιτικές και ότι έτσι είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει βιώσιμα η διαχείριση των δασών στην Ευρώπη. Άρα δεν πρέπει να σε το κριτήριο της βιωσιμότητας. πρέπει να ισχύει και για την ε, βιομάζα. Και αυτό βέβαια να ισχύει και για τις εισαγωγές από τις τρίτες χώρες. Και με τις ρυθμίσεις αυτές να βοηθήσουμε ε, διάφορες ε, κοινότητες και τις τρίτες χώρες να αναπτύξουν την ε, δασοκομεία και να μην έχουμε μεταξύ μας ε, ανταγωνισμό. Πολύ σημαντική βήμα για την ε, ευρωπαϊκή αγορά. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, λέει ο Πρόεδρος. Και, και τώρα. Όπως ακριβώς ζητήθηκε, ας ακούσουμε τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ρωτήθηκαν πολλά. Όλα αυτά που συζητήσαμε. Thank you, Chair. And thank you to... Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής που έθεσαν μια σειρά θερμα... θεμάτων για τη σημερινή συζήτηση. Σε αυτό το στάδιο, στην προπαρασκευαστική ε, φάση. Είναι δύσκολο να σας πω κάποια συγκεκριμένα πράγματα, γι' αυτό θα κάνω ελάχιστες παρατηρήσεις ε, που μπορώ να σχολιάσω. Να απαντήσω στο δικό σας ερώτημα, ε, κύριε Πρόεδρε, για τη βορρά εναλλαγής. Είναι, από ό,τι φαίνεται, ότι όταν κανείς κατά την αγρανάπαυση στην ουσία καλλιεργεί κάποια φυτά που ε, δεσμεύουν τον άνθρακο ε, είναι μια καλή τακτική για την αλλαγή του κλίματος ε, διότι με αυτόν τον τρόπο αυτά τα σπαρτά θα γίνουν μετά μια θετική συνεισφορά στη βιοενέργεια. Αν δούμε τον κατάλογο στο παράρτημα της οδηγίας Άλλοκ που αναφέρει ακριβώς αυτά τα... αυτές τις καλλιέργειες. Και υπάρχει και αυτή η πολιτική των αποβλήτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ε, ενέργειας, η αρχή κασκέτη των διαδοχικών χρήσεων, που στην ουσία δείχνει πόσο πιο αποδοτικοί μπορούμε να γίνουμε ε, όταν έχουμε αυτή τη χρήση των αποβλήτων, αντί να τα ρίχνουμε ε, στις χωματερές. Επίσης, ε, όσον αφορά στα κριτήρια βιωσιμότητας ε, πρέπει όσο ειδικά κι αν είναι ε, να έχουν αποτέλεσμα, να μην είναι απλώς ακριβή, διότι όταν κανείς στην ουσία φυτεύει ένα δέντρο, δεν μπορεί να ξέρει πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό 70-80 χρόνια μετά. Αυτό πρέπει να το διασφαλίσουμε και θέλουμε η πολιτική βιωσιμότητα να μην ε, έχει διακρίσεις εναντί τρίτων χωρών. Οι μελλοντικές ε, πολιτικές βιωσιμότητας ε, θα πρέπει να ενδιαφέρουν και τις άλλες χώρες, ώστε να την εισακολουθήσουν και αυτές. Επίσης, ε, η σωστή λογιστική, ο σωστός λογιστικός ε, απολογισμός της χρήσης της γης είναι κάτι που αναφέρθηκε. Όντως, ε, για να είμαστε ουδέτεροι ως προς την παραγωγή άνθρακα, είναι ε, πολύ σημαντικό να τηρήσουμε ε, σωστά λογιστικά στοιχεία, να γίνει σωστός υπολογισμός ε, και να συνάδει αυτός με τις υφιστάμενες οδηγίες του IPCC. Επίσης, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα επικουρικότητας, όπως αναφέραν πολλοί βουλευτές σήμερα. Και αν δούμε όλα αυτά τα στοιχεία ε, μέσα στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων για το κλίμα του 2030, μία από τις αρχές που θέλουμε να ακολουθήσουμε είναι η ευελιξία για τα κράτη-μέλη, τα οποία θα πρέπει αυτά να αποφασίσουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να επιτύχουν τους στόχους ε, στο τομέα των κτηρίων, της γεωργίας ή των μεταφορών. Και έτσι θα υπάρχει ε, μεγάλη ποικιλία στις ε, πηγές ε, που θα είναι διαθέσιμες στα κράτη-μέλη. Όμως πρέπει η βιοενεργία να χρησιμοποιείται και να αυξηθεί η χρήση της μέχρι το 2030. Πρέπει λοιπόν οι προμηθευτές και οι πελάτες να έχουν τη διασφάλιση ότι όλα αυτά θα γίνουν με βιώσιμο τρόπο. Η Κομισιόν Επίσης, θέλει να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές που θα προωθήσουμε ε, θα βοηθούν ε, στην διατήρηση μιας καλής ποιότητας αέρα. Ε, ότι δεν θα έχουμε στην ατμόσφαιρα σωματίδια τα οποία θα είναι βλαβερά και δεν θέλουμε ε, να περάσουμε σε μεγάλα ή μεσαία βεληνικούς εργοστάσια. Ε, αυτό το προσέχουμε ιδιαίτερα. Και μετά υπάρχει κι άλλο ένα θέμα που τέθηκε για την εντατικότητα της ενέργειας. Όντως, εξετάζουμε πόσο αποτελεσματικά μπορεί να καεί η βιομάζα σε σχέση με άλλες πηγές ενέργειας, διότι πολλές φορές χρησιμοποιούνται οι δασικοί πόροι με τρόπο λιγότερο αποτελεσματικό. Τουλάχιστον όταν καίγονται να μπορούν ε, να χρησιμοποιούνται με αποδοτικό τρόπο και να μπορούν να ανακυκλώνονται πολλές φορές. Θα σταματήσω εδώ κύριε Πρόεδρε και είμαστε στη διάθεση της Επιτροπής σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας, τις απαντήσεις. Και τώρα Κλείνουμε αυτό το θέμα και μπορούμε να ξεκινήσουμε με το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αλλά μάλλον να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα γιατί δεν είναι εδώ ο εισηγητής. Okay, five minutes of stop. Uh, Πέντε λεπτά διάλειμμα αναμένοντας τον εισηγητή. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να επανέλθουμε και να ξεκινήσουμε με το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η διάφορη αναθεώρηση της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοπικιλότητα. Δίνω αμέσως ε, ε, το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Ντέμες Μάκερ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στις 2 Φεβρουαρίου αυτό εδώ το Κοινοβούλιο ενέκρινε την ε, έκθεσή μου για την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα με μια στριπτική πλειοψηφία. Το Κοινοβούλιο λοιπόν έστειλε ένα μήνυμα τότε. Ένα σαφές ηχηρό μήνυμα προς την Κομισιόν και προς τα κράτη-μέλη χρειάζεται επιγόντως να παρθούν μέτρα σε υψηλό πολιτικό επίπεδο για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την απώλεια βεπικιλότητας. Την 1η Μαρτίου, μαζί με κάποιους συναδέλφους, έθεσε ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα αντιδράσει σε αυτή την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ζητήσαμε, παραδείγματος χάρη, μια καλύτερη εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας. Η απάντηση της Κομισιόν όχι μόνο έφτασε καθυστερημένα, αλλά ήταν εξαιρετικά ασαφής. Λέει η Κομισιόν, εξετάζουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να σεβαστούμε τις επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό τώρα παρέθεσα το τι μας απάντησε η Κομισιόν. Πέρα από το ασαφές της απάντησης, που είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, δεν δόθηκε καμία απάντηση για το αποτέλεσμα του fitness check. Το συζητούσαμε τις προάλλες με τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Τίμερμαντς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε μια συζήτηση έντονη, όπου ο κύριος Τίμερμαντς απλά έριχνε προπέτασμα καπνού, έτσι, πυροτεχνήματα. Εγώ ζητώ από τον κύριο Βέλα να κάνει ό,τι μπορεί, να πιέσει για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το ζήτημα. Και θέλω να υπογραμμίσω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας βρει σύμμαχους εφόσον ζητήσει οι στόχοι για τη στρατηγική βιοπικιλότητας να γίνουν σεβαστοί, να επιτευθούν. Η έκθεση για τη βιοποικιλότητα είναι μια έκθεση στρατηγικής αξίας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταστήσει ορισμένα, ορισμένα πράγματα σαφή. Ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση και δεν μπορούμε να χάσουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ και τώρα να δώσω το λόγο στον σκιώδη συγκεκριτή τον κύριο Λίντς. Συγγνώμη, δεν ήμουν έτοιμη. Α, όχι, ο κύριος Λίντς. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να πω κάτι που υπόθηκε από τον προλαλήσαντα διότι είναι η πρώτη συζήτηση για το θέμα της βιοπικιλότητας και τη στρατηγική βιοπικιλότητας, όπως επίσης και για το σχετικό θέμα του μη ανοίγματο της προστασίας της φύσης. Ε, να πω ότι έχω ενδιαφερθεί πολύ για το θέμα ε, που αναφέρει λεπτομερώς η Κομισιόν συγκεκριμένα το πώς ε, σε αυτό το νέο χρονοδιάγραμμα θα μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα. Τώρα που έχουμε ένα έγγραφο, στο οποίο υπάρχουν και τα πέντε κριτήρια της ε, στρατηγικής για την προστασία της φύσης που πληρούνται μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας ε, που θεσπίζονται με, στην στρατηγική για την προστασία της φύσης. Το γεγονός βέβαια ότι εκπληρώνονται τώρα αυτά τα κριτήρια ε, δεν ε, είναι δικαιολογία για να περάσουμε το θέμα το φθινόπωρο. υπάρχει ξεκάθαρα στην ανακοίνωση της Κομισιόν ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο ε, για πολλούς μήνες θα οδηγήσει τους συμμετέχοντες ε, στην εφαρμογή της οδηγίας σε αβεβαιότητα. Ε, αυτούς δηλαδή, που, δηλαδή στα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό θα ήταν καλό να έχουμε μια έτσι, ξεκάθαρη ανάγνωση. Ο κύριος Γκερμπάντη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Κομισιόν που είναι εδώ. Καλό θα ήταν να ακούσουμε πρώτα τη δήλωση της Κομισιόν και μετά να απαντήσουμε και να αντιδράσουμε. Να πω κάποια πράγματα που έχω παρατηρήσει. Συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές. Για μένα το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι πέρυσι ε, το λάβαμε μία έκθεση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, για την κατάσταση της φύσης και μετά τον Οκτώβριο είχαμε και την ανακοίνωση της Κομισιόν, τη δήλωση της Κομισιόν και στη συνέχεια έχουμε τώρα αυτή την ενδιάμεση αναθεώρηση που δείχνει ότι σε καμία περίπτωση δεν πετυχαίνουμε τους στόχους. Αυτό έχει να κάνει με την τάση και τις πιέσεις ε, στο οικοσύστημα. Έχουμε 14 ε, στοιχεία που πρέπει, 40 ε, στοιχεία που ε, θα πρέπει να μειωθούν ως προς την πίεση που ασκούν στα οικοσυστήματα και μόνο 7 έχουν πετύχει το στόχο. Τα υπόλοιπα 33 απλώς αυξάνουν, συνεχίζουν να αυξάνουν την πίεση. Έχουμε μεγάλη απόσταση λοιπόν από την επίτευξη των στόχων. Στο έγγραφο της Κομισιόν τον Οκτώβρη αυτά τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα. Άρα θα περίμενα μέχρι τώρα να υπάρχει μια στρατηγική διαχείρισης κρίσεων. Πώς αλλάζουμε αυτό το μοτίβο. Στη συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς είδαμε ότι συμφώνησε πλήρως με αυτή την ανάλυση και είπε και δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν προτάσεις για τη μετώπιση του ζητήματος. Το ερώτημό μου λοιπόν στην Κομισιόν είναι το εξής. Αύριο μεθαύριο, την επόμενη εβδομάδα, πότε μπορούμε να περιμένουμε τις προτάσεις της Επιτροπής για την Γεωργία, το κυνήγι, οτιδήποτε έχουμε που χρειάζεται για να έχουμε μία στρατηγική για τη βιοπικιλότητα που θα επιτύχει τους στόχους της, γιατί αν δεν κάνουμε τίποτα δεν θα πάμε πουθενά. Ευχαριστώ κυρία Χόκεν. Uh, <laughs> Denne gang vil jeg igen tale, dansk og Αυτή τη φορά, αυτή φορά θα μιλήσω δανεικά και ε, ενθαρρύνω τους Ολλανδούς ε, φίλους να μιλώ και αυτή τη γλώσσα του Ολλανδικά, διότι η μετάφραση είναι πολύ καλή. Από τα Ολλανδικά προς τα Δανέζικα τουλάχιστον. Πρέπει όλοι να το γνωρίζουμε αυτό. Ο κύριος Τίμερμανς κάθε φορά που έρχεται εδώ μας λέει όχι την τελευταία φορά όμως υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει να βελτιώσει τα πράγματα και ήταν σαφές ότι συμφώνησε ο κύριος Τίμερ μας μαζί μας ότι θα πρέπει να περάσει αυτό το μέτρο για να προχωρήσουμε και βέβαια χάρηκε ε, όταν εμείς τον επενέσαμε, όταν ε, ε, δείξαμε ότι τον καταλάβαμε και σήμερα από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος ακούμε ότι ε, η απάντηση είναι αρνητική και ότι αναμένονται βελτιώσεις. Βεβαίω είχε υποθεί από τον κ. κάποια στιγμή ότι αν κάτι δεν είναι, δεν είναι χαλασμένο δεν χρειάζεται να το φτιάξουμε αλλά στέλνουμε ένα μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Τίμερμανς μας έκανε μια υπόσχεση. Πρέπει να τηρηθεί, πρέπει να προχωρήσουμε. Μην αρχίζετε πάλι ε, να μας λέτε δικαιολογίες ότι υπάρχουν άλλα ζητήματα, το προσφυγικό, το ένα το άλλο. Αυτή η στρατηγική είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και στην εφαρμογή των κανόνων. Και όταν κάτι δεν πάει καλά με την εφαρμογή ε, των οδηγιών αυτών, ε, πρέπει να αντιδρούμε. Αυτές οι οδηγίες ε, έχουν τύχει πολύ θετική υποδοχή από τους συμπολίτε μας. πάντα τη χάνει καλή υποδοχή. Οποιαδήποτε διάταξη ενισχύει την προστασία της φύσης. Και κάτι ακόμα για την ανακοίνωση αυτή τώρα. Οι πολίτες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν εφόσον γίνει αυτή η ανακοίνωση. Η σύμβαση του άρχους που έχει να κάνει με τη συμμετοχή των πολιτών δεν είναι κάτι το οποίο το παίρνουμε αρκετά σοβαρά στο κοινοβούλιο αυτό. Έγινε μια συζήτηση ε, στην Επιτροπή Αναφορών για αυτήν την σύμβαση σήμερα και ξαφνικά ελέγχθη ότι δεν εφαρμοστεί η σύμβαση του άρχους σωστά. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα όμως. Εάν η Κομισιόν εκπονήσει την ανακοίνωση τώρα, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία τη σύμβασης του άρχους που να επιτρέπει τη συμμετοχή των πολιτών στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Αυτό θα μας βοηθήσει να σημειώσουμε πρόοδο σε μια χρονική στιγμή όπου πολλοί συμπολίτε μας ε, λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απόμακρη, είναι μη δημοκρατική. Είναι μια ευκαιρία να στείλουμε το κατάλληλο μήνυμα και αυτό είναι προς συμφέρον όλων. Και όπως ελέγχθη πολλές φορές, είναι αναγκαία η στρατηγική αυτή για να πετύχουμε τους στόχους μας για τη βιοπικιλότητα. Και ούτως ή άλλως ε, ήρθε η στιγμή να σημειώσουμε πρόοδο. Δεν μπορούμε συνεχώς να επαναχωρούμε. Και βλέπω ότι μόλις έφτασε και ο Καρλ Χάινς Φλόρενς, ε, και θα βοηθήσει και αυτός ελπίζω έτσι ώστε οι συμπολίτες μας συμμετάσχουν πιο ενεργά και θα έχουν τα καλύτερα εργαλεία στη διάθεσή τους για μια καλύτερη και πιο πράσινη Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριος Πότς, ευχαριστώ πρόεδρε. Εδώ έχω την ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής βιοποικιλότητας του 2020, έγγραφο που εκπώνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κάθε στόχος που αναφέρεται εδώ συνοδεύεται ε, από όρους όπως ανεπαρκής πρόοδος, ε, καμία ουσιαστική πρόοδος, ανεπαρκής, ε, καμία ουσιαστική ανεπαρκής. Ο μόνος θετικός στόχος είναι ο στόχος 5 για την καταπολέμηση των alien species. Να πω στην Κομισιόν ότι δεν τα πάτε καλά με την εφαρμογή, δεν ακολουθείτε το χρονοδιάγραμμα. Πρώτον, η Κομισιόν δεν σέβεται τον ίδιο τον κανονισμό. Δεν έχετε πράξη κατεξοδότηση για την αξιολόγηση κινδύνου. Δεν έχετε ένα κατάλογο ε, για τις, ε, τα alien species. Θέλετε να συμπεριλάβετε εδώ είδη τα οποία χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως, ε, στον τομέα της κτηνοτροφίας, ως ε, ζώα συντροφιάς, ε, τον βυσόνα, τον αμερικανικό υπάρχει και πρωτοβουλία, έτσι, να μπει στον κατάλογο ε, των ε, ειδών, ε, των εξωτικών ειδών των φυσικών των πολιτειών Ένα ζώο το οποίο υπάρχει σε ένα μόνο νησί και μάλιστα το 5% των μελετών λένε δεν υπάρχει. Και αυτό λέμε ότι είναι ένα εξωτικό ε, είδος το μόνο αποτέλεσμα των λεγόμενων προσπάθειών σας είναι ότι υπάρχει η αντίρρηση από το Κοινοβούλιο και, υπάρχει και αρνητική, αρνητικό ψήσμα του Ολλανδικού Κοινοβουλίου. Ε, δεν έχετε λοιπόν τίποτα και χάρη στην Κομισιόν, δυστυχώς, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτύχει για άλλη μια φορά με τους στόχους ε, για την επικοινότητα του 2020. Ευχαριστώ. Thank you Εμείς σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Τι τρώει το λόγο η κυρία Πύρικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Την ε, προηγουμένη εβδομάδα, εδώ, σε αυτή την ίδια αίθουσα, εξαντλητικά τα συζητήσαμε και δεν θα τα ξαναπώ. Αλλά μας είπε ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς ότι θέλει και αυτός να καθίσει το τι κάνει γιατί δεν κάνει η Ευρώπη, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει. Πολύ θετικό αυτό. Και έτσι μπορούμε καλύτερα να οριοθετήσουμε την ε, αξιολόγηση, την αναθεώρηση αυτήν που εγώ θα ήθελα να γίνει σε κάποιες οδηγίες και του τόπα και του εισηγητού στην παράγραφο 19 λέει ζήτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει ε, τις γραμμέ γραμμές όσον αφορά την εφαρμογή των οδηγιών, λαμβάνοντας υπόψη τα νομικά ζητήματα τα οποία ακόμη εκκρεμούν. Και επίσης ε, θα πρέπει να ενημερωθεί ο διάλογος μετα, μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής σε σε και όλων των εμπλεκομένων και ενδιαφερμένων και είναι πάρα πολύ σημαντική βέβαια οι κοινωνικοί παράγοντες. Να, περί τίνος πρόκειται και εγώ δεν είπα ότι πρέπει να γνωρίσουμε τις οδηγίες, αλλά κάποιοι είναι καλοί μαθητές και κάποιοι κακοί μαθητές. Εμείς κάναμε πολλά και με τις οδηγίες της βιοποικιλότητας γίνεται πολλή δουλειά στις διάφορες περιφέρειες. Για να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. κύριος ε, Φλόρεντ. Δεν ε, έχω και πολλά να πω τώρα, γιατί ε, έχω ήδη συζητήσει για το θέμα της εφαρμογής διαφορών κανόνων. Να μιλήσω μόνο για την διαχείριση των επιθετικών ειδών, που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν σκέφτομαι ε, πόσα τέτοια είδη έρχονται στο Αμβούργο μέσα από τα φορτία που έρχονται διαθαλάσσεις, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση. Η συνάδελφος Άουκεν, την οποία εκτιμώ ιδιαίτερα, να της πω κάτι. Όταν υπάρχει ε, ένα αν υπάρχει ένα μη δημοκρατικό εργαλείο είναι η σύμβαση ε, που ε, υπάρχει και ε, εντάξει υπάρχουν πολύ συμπαθητικοί κύριοι από τη χώρα σας που έχουν εμπλακεί σε αυτό, όμως χωρίς να υπάρχει κοινοβουλευτική κάλυψη αποφασίζουν κάτι και μετά λένε, λέμε ότι υπάρχουν στη σύμβαση και πρέπει να ισχύουν. Όταν δεν έχει αποφαστεί κάτι κοινοβουλευτικά, αν δεν υπάρχουν ε, συζητήσεις μεταξύ βουλευτών για τέτοια ζητήματα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι νομιμοποιούνται αυτά. Δεν πρέπει να είναι λοιπόν κάποιο μυστικό ανάγνωσμα αυτό που αποφασίζουμε, αλλά κάτι που συζητείται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Thank you much, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την παρουσίασή της. Νομίζω το θέμα της αποδοχής της Ευρώπης από τους πολίτες της, τους συμπολίτε μας, τίθεται ξεκάθαρα και αυτή η οδηγία που σε όλες τις χώρες δημιούργησε τεράστιες συζητήσεις συχνά είναι στο στόχαστρο ε, γιατί μιλά, η Ευρώπη στην ουσία ασχολείται με θέματα που θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν οι ε, τοπικές κοινωνίες. Νομίζω λοιπόν ότι ε, έχουμε περισσότερο υποχρέωση να έχουμε αποτελέσματα και όχι μέσα. Και τα κείμενα της Κομισιόν στην ουσία σέβονται αυτή την υποχρέωση για αποτελέσματα, επιτρέπουν στους ντόπιου να λαμβάνουν μέτρα τα οποία ε, θα είναι πιο προσαρμοσμένα στην ε, τρέχουσα κατάσταση εκεί και να μην ε, τα διαχειρίζεται κάποιος από μακριά. Λοιπόν, έχω εδώ κάποια νούμερα για το 2015 για το Λύκο και εκεί Έχουμε δώσει 15.800 ε, ευρώ για την προστασία του και έχουμε σχεδόν 9.000 θύματα ε, τα οποία πήραν 3 εκατομμύρια σε αποζημίαση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ε, πού βρισκόμαστε σήμερα. Πιστώσεις για προτεραιότητες που ορίζουμε καθημερινά όχι μόνο εδώ στην Επιτροπή αλλά και στην Ολομέλεια και στην ομάδα θα πρέπει η Ευρώπη να είναι πιο ρεαλίστρια στις πολιτικές της, νομίζω. Thank you very much. If, uh, no Κύριε Άουκεν ζήτησε, ναι, για τον Κάρλ Χάινς να του πω πολύ σύντομα ότι το 2006 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε μία νομοθετική έκθεση η οποία ε, μιλούσε για αυτή τη σύμβαση η οποία ε, ήταν αντικείμενο μεγάλη συζήτηση, ε, ήταν πολύ δημοκρατική αυτή η συζήτηση, ακόμα και αν δεν σας αρέσουν οι άνθρωποι που είναι στη δικιά σας αυλή, συζητήθηκε δημοκρατικά, εφαρμόστηκε, αλλά δεν χρησιμοποιείται. Και ο Μπίλαντ σήμερα είπε ότι είναι κατά της διαφάνειας, ήρθε πέντε λεπτά πριν κλείσουμε σήκωσε το χέρι και είπε είμαι κατά. Αυτό ήταν σκάνδαλο. Η μάνα του θα ντρεπόταν. Όμως έχει συζητηθεί αυτή η σύμβαση και είναι η βάση για τη συμμετοχή των πολιτών. Simply wrong, ε, κάνετε λάθος, αλλά εντάξει. Αν σταματήσουμε τη συζήτηση εδώ μεταξύ μας. Καλύτερα να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια θα καλέσω τον κύριο Ρόζα για να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα αλλά και να μας αναφέρει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ε, κύριε Συγητά, αξιότιμα μέλη φαίνεται εδώ ότι το Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να παίξει ένα κεντρικό ρόλο για να προστατεύσει το φυσικό κεφάλαιο της Ένωσης. Είναι επίση μια ευκαιρία εδώ να διακρινούμε κάποια σημεία για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το σημαντικό έργο, μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση ε, για τη βιοπικιλότητα και την ψήφιση του Κοινοβουλίου. Είμαι έτοιμος να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα και να τονίσουμε και το ρόλο που παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία. Ξεκινώντα ε, με την οδηγία να πω ότι η Κομισιόν υποστηρίζει τους κανόνες για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ξέρετε, κάναμε μια μεγάλη ανάλυση στοιχειοθετημένη τα πρώτα ευρήματα της σχετικής έκθεσης έχουν δημοσιοποιηθεί από τον Νοέμβριο. Η πλήρης έκθεση θα είναι διαθέσιμη από κοινού με, τη με το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ιστορική διαδικασία της Κομισιόν δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να επανέλθει στο θέμα αυτό το φθινόπωρο, να παρουσιάσει ε, τα αποτέλεσμα του fitness check μαζί με κάποιες δράσεις follow-up. Δεν έχουμε σταματήσει όμως, συνεχίζουμε την εφαρμογή και την παρακολούθηση ε, των οδηγιών συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για την προώθηση ε, της συντήρησης και της βιώσιμης χρήσης του Natura 2000 ε, προς ε, όφελος της φύσης και των ανθρώπων. Όταν προκύπτουν προβλήματα, διενεργούμε έρευνα και όποτε χρειαστεί παρεμβαίνουμε και νομικά. Πρόσφατα, την περσμένη εβδομάδα, ε, πήραμε απόφαση για διαδικασία που παραβάσει σε ό,τι φορά την οδηγία ε, για το ε, υγροβιότοπο για τους βιοτόπους μάλλον. Το πρασίνισμα στην, στις, στις πληρωμές του πρώτου πυλώνα στον τομέα της γεωργικής πολιτικής μας δίνει τη δυνατότητα να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του πρασινίσματος στα πλαίσια επικοινότητας μειώνοντας το διοικητικό άχθος. Ένα έγγραφο εργασιών θα παρουσιαστεί σύντομα για να καταδείξει οδούς απλοποίησης και βελτίωση των διατάξεων περί πρασινίσματο και καλό θα είναι να έχουμε την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό, καθώ και για την ενδεχόμενη αύξηση ε, των υποχρεωτικών ε, τη υποχρεωτική γη για βιολογικού σκοπού από το 5% στο 20%. πρέπει να παρακολουθούμε την αναθεώρηση του πρασινίσματο, ε, τα αποτελέσματα των προγραμμάτων ανάπτυξη υπαίθρου και να χρησιμοποιήσει τι δυνατότητε που έχει για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει πολιτική εφαρμογή. Σε Ό,τι αφορά την προστασία ε, των υγροβιότοπων, των οικοσυστημάτων μάλλον, των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, πλησιάζει η αξιολόγηση. Θα μπορέσουμε να δούμε κατά πόσο τα κράτη-μέλη και η στρατηγική ε, για το θαλάσσιο περιβάλλον προχωράει καλά. Πρόσφατες μελέτες ε, θα μας βοηθήσουν να βρούμε τους καλύτερους τρόπους για να προωθήσουμε τις πράσινες υποδομές και να μειώσουμε ε, την απώλεια βιοποικιλότητας πέρα από το Natura 2000. Επίσης, γίνονται εργασίες για το Natural Capital Accounting σε ό,τι αφορά τα χωροκατακτητικά είδη. Σύντομα θα έχουμε μια ανακοίνωση της Κομισιόν, θα συνεχιστούν και εξολογήσεις κινδύνου και για να απαντήσω στις κριτικές που ακούστηκαν ε, για τα ήδη αυτά. Ε, το πρώτο σχέδιο καταλόγου για τα ίδια αυτά βασίστηκε σε μια συστηματική και επιστημονική προσέγγιση χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες αξιολογίες κινδύνου και συμμορφόμενοι με ε, τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού για τα χωροπρακτικά ε, ξένα ε, Βασιζόμαστε λοιπόν στα κριτήρια που υπάρχουν στον ίδιο το κανονισμό. Δεν έχουμε συμπεριλάβει λοιπόν εδώ κάποια είδη, ε, όταν δεν έχουν συμπληρωθεί κάποια είδη, είναι, είτε επειδή δεν συμμορφωνόντουσαν με τα κριτήρια, είτε επειδή δεν λέφθησαν υπόψη άλλα αριθμιστικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη σχέση κόστους-οφέλους των μέτρων. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα προβληματικά είδη τα οποία πρέπει να εξεταστούν. Γι' αυτό αρχίσαμε τα, τις νέες αξιολογήσεις ε, κινδύνου για τη μελλοντική επικαιροποίηση του καταλόγου και ο κατάλογο αυτό θα επικαιροποιείται όπως άλλωστε θα απαιτείται από τον κανονισμό. Επίσης πρόσφατα εγκρίναμε το σχέδιο δράσης για, για τη wildlife και λαμβάνει η χώρα και μία μελέτη για, τις, για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ξέρετε, πολλά από αυτά τα, τα θέματα συνδέονται άμεσα ή έμεσα με τη βιοπικιλότητα. Για να πετύχουμε του στόχου τη βιοπικιλότητα, πρέπει βεβαίω να μα υποστηρίξουν ευρύτερε πολιτικέ πρωτοβουλίε, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, παραδείγματο χάρη, ε, κάποια δικλείδα ασφαλεία για το κράτο δικαίου και πτυχέ ε, που έχουν να κάνουν με το κόστο. Η πρωτοβουλία για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη το 2016, ε, συμβουλή για τις υποθέσει που πάνε στο δικαστήριο, όλα αυτά πρέπει να τα μπορεί να τα παρέχει ένα κράτο μέλο. Ε, τέλος, ε, η διαδικασία για την περιβαλλοντική εφαρμογή θα υποστηρίξει την εφαρμογή της υπάρχους, των υπάρχων περιβαλλοντικών κανόνων και δεσμεύσεων και θα ακολουθήσει και κακολούθως μετά την έγκριση της EAR ε, τον περασμένο μήνα 28 εκθέσεις κρατών μελών έχουν προετοιμαστεί αλλά ε, αναφέροντας στα κενά στην εφαρμογή αλλά και τι βέλτιστες πρακτικέ με ειδική αναφορά στη βιοπικιλότητα. Η έκθεση θα καλύπτει την πολιτική τη νομικές δεσμεύσεις στην τομέα τη περιβαλλοντική πολιτικής, καθώς και την κυκλική οικονομία, τα απόβλητα, την ε, ρήπανση τη θάλασσα, την ατμοσφαιρική ρήπανση, τη βιοπικιλότητα όπω είπα και θα συνοδεύεται αυτό από συζητήσει ε, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κτλ. Θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε τα αιτήματα για νομοθετικέ πρωτοβουλίε που προκύπτουν από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως η έκκληση να λάβουμε δράση για τους pollinators, θα έχουμε τη δυνατότητα να το, να συζητήσουμε αυτό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του εμπλεκόμενου φορεί να βρούμε τον πιο κατάλληλο τρόπο για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Please, if you want to add something. Έχετε το λόγο αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Εγώ, Πρόεδρε, ήθελα όχι να προσθέσω κάτι. Απλώς ελπίζω επιτέλους. Α, μου απαντήσει η Επιτροπή στην ε, ερώτησή μου. Την έχω υποβάλει τέσσερις φορές, ούτε μία ούτε δύο. Το ίδιο πράγμα. Είναι θεμητό να το ρωτάει κανείς αυτό το πράγμα. Τι γίνεται με την ε, προσαρμογή των ε, ε, καθεντηρίων γραμμών που έχουμε ζητήσει με το ψήφισμά μα. Σα είπα ότι οι διοικητικέ περιφέρειε στην Ολλανδία ε, μερικέ τα, τα τηρούν, μερικέ όχι. Τι θα γίνει, θα προσαχθούν να πούν το δικαστήριο επί παραβάση. Τι γίνεται τώρα με τι χώρε που, που, που είναι καλοί μαθητέ και με αυτού που είναι κακοί μαθητέ. Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα 100% μιλάτε για την ε, εφαρμογή του Natura 2000 και του Regio. Φυσικά και συνεργάζομαι το κράτη μελή όσον αφορά την εφαρμογή των ε, ε, κρατών μελών. Και έχουμε επίσης τις σχετικές ε, εκθέσεις και εστιάζουμε προσοχή μας σε αυτές τις οδηγίες. Άρα συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για το θέμα τη εφαρμογή των οδηγιών. Δεν ξέρω μήπω ε, αναφέρεστε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο που αφορά την ε, ε, ε εφαρμογή. Εάν ξέρω να σας πω. Η συγκεκριμένη μου ερώτηση ήταν η εξή. Εκπονείται τώρα κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ, guidelines, στις κάτω χώρες, στην Ολλανδία, σε κάποιες περιφέρειες όπως η Χέλτερλαντ έχουν προχωρήσει πολύ όσον αφορά την υλοποίηση, την εφαρμογή. Έρχονται επομένω οι βουλευτέ των Περιφερειακών Κοινοβουλίων και μα λένε ότι δεν έχουν πολύ περιθώριο ενέργεια γιατί δεν έχουν τι κατευθυντήριες από πλευρά τη Ευρώπη. Εσεί πώ το βλέπετε, για να ξέρω και εγώ τι θα πω στην εκλογική μου περιφέρεια. Επιτροπή. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε δώσει κατευθυντήριες για διάφορες πτυχές των ε, οδηγιών, ούτω ώστε να μπορέσουν κάποιες κοινωνικές δραστηριότητε να είναι συμβατές με τις ε, οδηγίες. Ιχθυοκαλλιέργειες, δασοπονία κλπ. Σε διάφορες δραστηριότητε. Ίσως αυτό δεν αργεί, αλλά Το fitness check προέκυψε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η καθοδήγηση. Χρειάζεται. Συμφωνούμε ότι είναι σημαντικό και θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε και να δίνουμε κατευθυντήριες όπου χρειάζεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Και τώρα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, ο κ. Ντεμέης Μάγκερ που είναι ο συγητής. Πρόεδρε. Μου επιβεβαιώθηκε, μα βεβαίωσε η Κομισιόν ότι τα αποτελέσματα του fitness check θα τα λάβουμε το φθινόπωρο. Αυτό μας είπε η Κομισιόν. Εμείς δεν είπαμε ότι η Κομισιόν δεν κάνει τίποτα εντωμεταξύ. Έχουμε ένα πλήρη κατάλογο του τι κάνει η Κομισιόν. Όμως, κατά κάποιο τρόπο αποφύγατε το ερώτημά μου. Εγώ ρώτησα γιατί αυτή η καθυστέρηση η επίσημη απάντηση είναι ότι είναι η κρίση των προσφύγων στη μέση και ότι αυτό ε, μας οδηγεί στο έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη πρόκληση και ότι η Κομισιόν δεν μπορεί να προετοιμάσει ε, το έγγραφο. Ακούστε, μου φαίνεται κάπως φτηνή δικαιολογία αυτή. Σε τι οφείλεται λοιπόν αυτή η καθυστέρηση. Από πλευράς τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής από πλευράς ε, κρατών μελών ε, φαίνεται να υπάρχει βούληση να προχωρήσουμε. Οι οδηγίες πρέπει να είναι fit for purpose, βεβαίως. Όμως υπάρχουν καθυστερήσεις. Και εγώ δεν μπορώ παρά να εικάσω γιατί υπάρχει καθυστέρηση. Υπάρχει υποστήριξη Υπάρχει υποστήριξη ευρεία για αυτές τις οδηγίες. Τι περιμένει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε δίκιο, το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να παίζει ένα σημαντικό κεντρικό ρόλο για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε το, το φυσικό μας κεφάλαιο με μεγάλο πάθος να το υπερασπιστούμε μάλιστα. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Θέλ, θέλετε, περιμένετε απάντηση από την Κομισιόν. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ για το ερώτημα. Νομίζω ότι μπορώ να εξηγήσω. Ε, βεβαίως, μία πτυχή, ένα θέμα είναι το fitness check και τα ευρήματά του και τα συμπεράσματα από τα οποία θα πληθούν από εκεί. Αλλά θέλουμε να, να έχουμε και δράσεις. Το follow-up δηλαδή αυτού του fitness check. Και θα χρειαστεί χρόνος να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε ποιες δράσεις θα προτείνουμε. Αυτό είναι που εξηγεί το ότι θα έρθουμε ξανά το φθινόπωρο. Διότι το φθινόπωρο δεν θα έχουμε μόνο το fitness check, θα έχουμε και τις δράσεις που θα ακολουθήσουν το fitness check. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μπορούμε να κλείσουμε εδώ τη συζήτηση. Να σας θυμίσω ότι η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής ΕΝΒΗ θα γίνει στις 11 Ιουλίου. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Καλό σας βράδυ.